Uh, have probably uh, noticed, today is the e Ξέρετε ότι σήμερα είναι η μέρα εναντίον του τράφικινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τιμή που προεδρεύω σήμερα με τον συναδέλφο Πιμέντα Λόπες, αντιπρόεδρο της Επιτροπής ε, Γυναικείων Υποθέσεων και Ισότητας των Φύλων και να καλωσορίσω και τον Επίτροπο κύριο Αβραμόπουλο όταν έρθει. Το θέμα το έθεσαν στην ημερήσια διάταξη οι συντονιστές και αυτό είναι πάρα πολύ εύθετο. Το τράφικινγκ είναι μια σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 2011 Ξεκινήσαμε λοιπόν με την οδηγία εναντίον του τράφικινγκ. Ενισχύθηκε με περαιτέρω ρυθμίσεις το 2016 και το 2017. Περιλαμβάνονται μέτρα για μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Να υπενθυμίσω ένα μόνο πράγμα, την σημασία εφαρμογής ε, των μέτρων της οδηγίας αυτής για να καταπολεμηθεί η ατιμορρησία. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ επανειλημμένα έχει ζητήσει από τα κράτη-μέλη να ποινικοποιηθούν ε, κάποιες ενέργειες, ε, ε, κάτι το οποίο δεν γίνεται με απόλυτο τρόπο σήμερα. Την προηγούμενη φορά τα είχαμε συζητήσει όλα αυτά στα πλαίσια μιας κοινή ε, ε, ακρόασης για το τράφικινγκ γυναικών και παιδιών, στα πλαίσια της ε, μεταναστευτών, μεταναστευτικών φαινομένων και των προσφυγικών φαινομένων. Θα πρέπει και το 2018 λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να μείνουμε στα λόγια. Και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει μόνο τους πρόσφυγες, αλλά και πολλούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να κατανοήσουμε πώς οργανώνεται και διεξάγεται το τράφικινγκ. Πριν το τέλος του χρόνου περιμένουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 23, όπως και την έκθεση προόδου σύμφωνα με το άρθρο 20, η συνάντηση σήμερα έχει σαν στόχο την εκκίνηση εφαρμογής ειδικών μέτρων ε, ε, με την ενσωματωμένη προβληματική του φύλου. Η μελέτη έχει γίνει από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων. Πριν δώσω το λόγο στους ε, φιλοξενούμενους ομιλητές μας, θα ήθελα να ζητήσω από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών να κάνει μια μικρή εισαγωγή. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Ευχαριστώ όλους τους παριστάμενους. Σας ευχαριστώ που σε αυτή την ακρόαση μου επιτρέπετε να θέσω το θέμα της σωματεμπορίας και του λαθρεμπορίου ανθρώπων. Το θέμα της σωματεμπορίας συνδέεται σαφώς με το οργανωμένο έγκλημα. Και ξέρουμε πολύ καλά τις, στρατηγικές, ε, τις εκβιαστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται, κυρίως απέναντι στις γυναίκες και στα παιδιά. Συχνά και εναντίον ανδρών, ε, που προέρχονται όμως από πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Η Επιτροπή Γυναικών κατ' επανάληψη έχει εγγύψει του θέματος και έχουμε τονίσει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά πέφτουν δυσανάλογα θύματα στα πλαίσια αυτού του φαινομένου. Και το φαινόμενο αυτό της αιμοτεμπορίας είναι μία μορφή βίας κατά των γυναικών. Και τροφοδοτεί και την σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών ένα άλλο άθλιο εμπόριο. Πριν έρθω εδώ στην ε, ακρόαση, προσπάθησα να βρω κάποιες πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ιστοσελίδα της δίνει κάποιες πληροφορίες, οι οποίες μοιάζουν όμως αντιφατικές. Βρήκα μια πληροφορία ότι περίπου 80% των θυμάτων σωματεμπορίας προορίζονται για σεξουαλική εκμετάλλευση. Έχουμε 18% καταναγκαστικής εργασίας ή αναγκαστικής εργασίας. Ενώ αλλού μιλάμε για το 70% των ανθρώπων που πέφτουν θύματα σωματεμπορίας που προορίζονται για καταναγκαστική εργασία. Εμείς πιστεύουμε περισσότερο στα πρώτα νούμερα αυτά, 80-18 δηλαδή. Ότι η μεγάλη πλειοψηφία δηλαδή των ατόμων αυτών την χάνουν εκμετάλλευση και βρίσκονται και καταλήγουν στα δίκτυα πορνείας. 95% των γυναικών που πέφτουν θύματα σωματεμπορίας και που είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης είναι γυναίκες. Τα πρόσωπα αυτά είναι κυρίως γυναίκες. Όμως υπάρχει και μεγάλη σχέση ανάμεσα στη σωματεμπορία και στα ναρκωτικά. Δηλαδή μέσω ε, αυτού του φαινομένου στην πραγματικότητα ξεπλύνουμε προσόδους από άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Πιστεύουμε ότι αυτή η συζήτηση για τη σεξουαλική εκμετάλλευση στα πλαίσια της σωματεμπορίας, στα πλαίσια του λαθρεμπορίου ανθρώπων και οι απαντήσεις που δίνουν τα κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η σεξουαλική εκμετάλλευση και γενικά η πορνεία θα πρέπει να μας απασχολήσουν πάρα πολύ και να δώσουμε απαντήσεις στο φαινόμενο της, του λαθρεμπορίου ανθρώπων. Ε, επίσης υπάρχει σχέση ανάμεσα στην αύξηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και στη σωματεμπορία. Γιατί τα πρώτα φαινόμενα αυτά, ε, η φτώχεια λοιπά, ε, καθιστά πιο ευάλωτα διάφορα στρώματα, διάφορες γυναίκες και τελικά πέφτουν θύματα σωματεμπορίας. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ε, δημιουργούνται οι συνθήκες για ένα τέτοιο φαινόμενο. Σας ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσε αρχικές παρατηρήσεις και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μαρία Μύρια Βασιλιάδου, που είναι η συντονίστρια τη Ευρωπαϊκής Ένωση κατά του φαινομένου της σωματεμπορία. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ και τους Προέδρους των δύο Επιτροπών ε, για την διάθεσή τους να συνεργαστούν για το θέμα αυτό η δουλειά του Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ φιλόδοξη και σας καλωσορίζω όλους σε αυτήν την ακρόαση ε, θερμά. Είναι η 12η ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολέμησης της ε, σωματεμπορίας. Υπάρχουν χιλιάδες άντρες και γυναίκες που πουλούνται, αγοράζονται και πουλούνται στην αγορά προς ε, εκμετάλλευση και για το κέρδος. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να θυμηθούμε επίσης ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια πολύ σοβαρή μορφή οργανωμένου εγκλήματος που είναι και παραβίαση ταυτόχρονα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων για τη δουλειά που κάνουν προς αυτήν την κατεύθυνση, για την έκθεσή τους και όλα αυτά δείχνουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε, τη δουλειά που κάνουμε με την υπογραφή της κοινή δήλωση μεταξύ 10 οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συνεργαστούμε για να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο της σωματεμπορίας. Ε, η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Διάστασης ε, για να δοθεί μια προοπτική φύλου ε, στο θέμα του trafficking ε, και είπαμε από το 2016 ότι είναι ε, διαρθωτική βία εναντίον των γυναικών και των κοριτσιών. Και η οδηγία κατά του τράφικινγκ ε, δημιουργεί νομικέ υποχρεώσει προ τα κάτι μέλη να υιοθετήσουν μέτρα τα οποία είναι συγκεκριμένα για το φύλλο. Δεν είναι ιδεολογικό το θέμα, είναι νομική υποχρέωση που έχουν τα κράτη-μέλη. Απορρέει, ε, ξεκινάει με την δημιουργία ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και προσπαθούμε να αποτρέψουμε αυτό το έγκλημα. Και αυτό αντανακλάται στην ανακοίνωση του 17 μας και στις προτεραιότητες που παρουσιάσαμε στο Κοινοβούλιο ήδη και σε παλιές εμφανίσεις. Το 2016 ξεκινήσαμε μια μελέτη για την ε, διάσταση του φύλου στα πλαίσια του λαθρεμπορίου που δείχνει ότι η βοήθεια προς, τους, ε, προς τα θύματα ε, από τη βοήθεια που δίνουμε ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με το φύλλο αυτή η διάσταση. Είναι πολύ σοβαρές, μακροπρόθεσμες αυτές οι ζημιές ε, γυναικολογικές, ψυχολογικές ε, και μπορεί να δημιουργήσουν τραύματα διαβίου μόνο και μόνο για να τις εκμεταλλευτούν ε, σεξουαλικά αυτές τις γυναίκες και κορίτσια. Ε, γι' αυτό λοιπόν το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι η νομοθεσία αυτή να λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου. Και νομίζω ότι το κάνει αυτό και ελπίζω το κάνει η έκθεση. Ευχαριστώ την πρόεδρο που μίλησε για τα, τον πρόεδρο που μίλησε για τα δεδομένα. 67% των θυμάτων ε, το 2014 ήταν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και η συντριπτική πλειοψηφία ήταν κορίτσια και γυναίκες. Ε, η Κομισιόν στο τέλος του 2018 θα έχει και συγκεκριμένα δεδομένα για τα καταχωρημένα θύματα, όχι απλώς για τις εκτιμήσεις, για τις μορφές εκμετάλλευσης, αλλά είναι αναφυσβήτητο ότι πρόκειται για έγκλημα το οποίο κυρίως επηρεάζει τις γυναίκες και τα κορίτσια. Επίση, ξέρουμε ότι έχουμε όλο και περισσότερε γυναίκε και κορίτσια που διακινούνται για λόγου σεξουαλική ε, εκμετάλλευση μέσω παρανόμων διόδων ε, μετανάστευση. Ε, η κεντρική με, Μεσόγειο. Ε, έχουμε 600% αύξηση από το 2014 αυτών των ροών και αυτό συνάδει με τα απορίσματα της Frontex το 2018 είναι αναφυσβήτα αυτά τα στοιχεία. Ε, δυστυχώς, βλέπουμε όλο και λιγότερο ε, να διακινούνται άτομα α, ή μάλλον να αντιμετωπίζει το θέμα της α, σωματεμπορίας ε, για λόγους σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Επομένως, είμαι πολύ ευγνώμων προς το Κοινοβούλιο που εξασφαλίζει την εστίαση στα, στις ανάγκες των θυμάτων και ούτως ώστε να μην τα περιθωριοποιήσουμε δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι μπορέσαμε να μειώσουμε την ε, επίπτωση του φαινομένου του trafficking για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ξέρουμε ότι τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα είναι όλο και πιο ευέλικτα και βρίσκουν νέους τρόπους ε, για να προσελκύσουν θύματα. Η Χιροπόλ λέει ότι η συνεχή ζήτηση για υπηρεσίες που συνδέονται με την εκμετάλλευση και οι πολύ μεγάλες ανισότητες ανάμεσα στον αναπτυγμένο και στον αναπτυσσόμενο ε, κόσμο ε, αυξάνουν τη ζήτηση. Δεν το λέω εγώ αυτά, τα λέει η Europol. Και λέει ότι υπάρχουν κράτη-μέλη όπου η πορνεία είναι νόμιμη και γι' αυτό οι διακινητέ ε, έχουν εύκολου δρόμου για να χρησιμοποιήσουν νόμιμε οδού για να εκμεταλλευτούν τα θύματα του. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα θύματα τα εντοπίζουμε και έχουν πρόσβαση σε βοήθεια και σε στήριξη. Δυστυχώ, ξέρουμε από την αναθεώρηση τη πολιτική μα ότι όταν η Κομισιόν δημοσίευσε όλα τα project ε, που χρηματοδοτήσαμε το 2003 μέχρι σήμερα, εκτός από την κρίση της μετανάστευσης, ξέρουμε ότι η μέση χρηματοδότηση ανά project για την εκμετάλλευση εργατικού δυναμικού ε, ήταν διπλάσιο ε, για θέματα ε, εκμετάλλευσης της εργασίας. Αλλά πάντα ξέρουμε ε, ότι βρίσκουμε αυτό που ψάχνουμε. Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε ποτέ να ψάχνουμε ποια είναι αυτά τα θύματα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ε, εύκολα μπορούμε να πούμε ότι η σωματεμπορία ε, συμβαίνει γιατί ο κόσμος είναι ευάλωτος. Εύκολα να το πεις. Ε, δεν συμβαίνει γι' αυτό όμως. Δεν συμβαίνει. Συμβαίνει γιατί υπάρχει το κέρδος, υπάρχει το χρήμα από πίσω. Και συμβαίνει γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τα σημεία ε, του ευάλωτου ανθρώπου. Αν δεν υπάρχει ε, κέρδος, αν δεν υπάρχει χρήμα, αν δεν υπάρχουν διακινητές, ε, δεν υπάρχει ε, σωματεμπορία. Η Europol ε, δημοσίευσε από μισή ώρα μια έκθεση για την σωματεμπορία παιδιών που λέει ότι η διακίνηση ανηλίκων για σεξουαλική εκμετάλλευση είναι πολύ επικερδής. Ακούστε το, σήμερα υπόθηκε αυτό, γιατί οι εγκληματίες ξέρουν ότι οι πελάτες τους ονομάζουν ε, πελάτες, εγώ τους ονομάζω βιαστές. Είναι έτοιμοι να πληρώσουν περισσότερα για σεξουαλικές συναντήσεις με ανήλικους από ότι με ενήλικους. Ε, αυτό σημαίνει ότι οι βιαστές ε, ενδιαφέρονται για παιδιά και πληρώνουν και πολύ περισσότερα από ότι για ενήλικες. Τα λέει η έκθεση αυτή που εκδόθηκε πριν από μισή ώρα. Κάποια από τα κορίτσια είναι 7 χρονών. 6-7 χρονών. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντική και σημαδιακή αυτή η μέρα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είσαι σήμερα εδώ. Ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη ζήτηση γιατί είναι νομική υποχρέωση. Πρέπει να προλάβουμε το έγκλημα γιατί είναι ηθική και νομική υποχρέωση να το κάνουμε. Και ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε είναι να σταματήσουμε αυτή την κουλτούρα ατιμορρησίας. Αυτό που συμβαίνει όταν βιαστεί ένα 7χρονο κορίτσι από ένα βιαστή που πλήρωσε πολλά λεφτά. Ε, είναι ότι ο τύπος αυτός είναι εξαφανισμένος. Πού είναι αυτός ο τύπος. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κουλτούρα τιμωρησία. Όπω είπε η Κομισιόν το 2016, σε πολλά κράτη-μέλη δεν είναι παράνομο να χρησιμοποιήσουμε ή να αγοράσουμε υπηρεσίε ε, ε, ενό ανθρώπου που θα μα εξυπηρετήσει ε, ε, σεξουαλικά και είναι θύμα ε, trafficking. Είναι ε, υποχρέωση και προτεραιότητα της Κομισιόν να αντιμετωπίσει τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να ποινικοποιήσουν αυτό το φαινόμενο ε, και να τιμωρήσει αυτούς που χρησιμοποιούν τέτοιες υπηρεσίες. Θα ήθελα να σας πω, έχετε δει ποτέ Μερικοί, μερικοί ισχυρίζονται ότι δεν κατάλαβαν, ότι δεν ξέραν πόσο χρονών είναι κτλ. Έχετε δει ποτέ εφτάχνο κορίτσι που δεν έχετε καταλάβει πόσο νεαρό είναι. Είναι απαράδεικτο να θεωρούμε δεδομένο ότι κάποιο ο οποίο είναι ευάλωτο είναι λογικό να πέσει θύμα. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή, σε ένα σημείο που να λέμε: Οκ, okay, τα εκμεταλλευόμαστε, τα διακινούμε αυτά τα άτομα και περιμένουμε ότι η αδυναμία του σημαίνει κατά ανάγκη και τη θυματοποίησή τους. Θα πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή τη λογική, αυτή την και θα πρέπει όσοι κερδοφορούν από αυτή την, ε, αυτό το φαινόμενο, όσοι αγοράζουν τέτοιες υπηρεσίες, πελάτες αυτών των προϊόντων, χρήστες. Και όλους όσους καταχρώνται αυτά τα άτομα, όλοι αυτοί θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Και πώς να θα λογοδοτήσουν, αν υπάρχει δίκαιο. Θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τι πράξει τους. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε αυτή την έκθεση. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία για να εφαρμόσουμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για το τράφικινγκ. Ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο για αυτό το ευρύτατο εργαλείο και είναι απαράδεκτο να μην βάλουμε και τη διάσταση του φύλου. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε, το λένε όλοι οι δείκτες. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Βασιλιάδου για τα λόγια σας. Η κυρία Βεζνή Ντελαμπάκ έχει το λόγο από το Ινστιτούτο Ισότητας των Φίλων. Ευχαριστώ. Ακούγοντας τα στοιχεία, σκεφτόμουν ότι σήμερα, αύριο, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει κίνδυνος κάποιος από εμά να μην βρει την αδερφή του, την κόρη του, ε, τη φοιτήτριά του και δεν θα ξέρουμε πού θα είναι, δεν ξέρουμε τι θα της έχει συμβεί, δεν ξέρουμε πότε θα την ξαναδούμε, αν θα την ξαναδούμε. Και στην σημερινή ψηφιακή εποχή Βλέπουμε ολοένα και περισσότερα κυβερνοεγκλήματα, τρόποι που αξιοποιούν το διαδίκτυο για να παγιδεύονται κορίτσια ε, και να οδηγούνται σε επικίνδυνους δρόμους. Γι' αυτό και όπως ε, υπόθηκε χρειάζεται να, να δημιουργήσουμε και να διαμορφώσουμε νέα μέτρα. Γιατί οι κίνδυνοι δεν μειώνονται, αυξάνονται και όπως υπόθηκε το 95% των θυμάτων του τράφικινγκ είναι γυναίκες και κορίτσια. Και δυστυχώς αυξάνεται και το ποσοστό των ανηλίκων μεταξύ των θυμάτων. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικά τα στοιχεία αυτά. Βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο γύρο ε, για την καταπολέμηση του τράφικινγκ της διαδικασίας της επίσημης που έχει θεσπιστεί και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η έκθεση που συντάξαμε ακριβώς για να αναδείξουμε τη διάσταση του φύλου που συνδέεται με την ανισότητα, με, τις, με, την, με, τις, με την εξουσία που ασκείται ε, εις βάρος των γυναικών τη βία που ασκείται εις βάρος των ε, γυναικών. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε εμείς από τη δική μας πλευρά. Βεβαίως η, η Ευρωπόλ έχει άλλο καθήκον να δει τα εγκληματικά στοιχεία. Εμείς όμως το καθήκον μας είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα μέτρα που λαμβάνονται για να βελτιωθεί η κατάσταση, για να, μειωθεί, για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο του τράφικινγκ. Και στην έκθεσή μας ε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει όλοι οι φορεί να αλληλοσυμπληρώνονται οι δραστηριότητες τους, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις Βεβαίω, η οδηγία για την κατολέμηση του τράφικινγκ ε, ξεκαθαρίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα του κάθε εμπλεκόμενου. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των κρατών μελών, υπάρχουν συγκεκριμένε αρμόδιες αρχές που προβλέπονται από την οδηγία. Επίσης η οδηγία ε, απαιτεί τη συμμετοχή των υποστηρικτικών οργανώσεων και το ξέρουμε όλοι ότι οι οργανώσεις γυναικών, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι εκείνες που έχουν τις γνώσεις που δεν έχουν συνήθως οι επίσημες αρχές και βοηθούν πολύ στην κατανόηση γιατί μία από τις διαστάσεις που αναφέρθηκε σήμερα και από τους προλαλήσαντες σχετίζεται με την ανισότητα των φίλων βεβαίως, αλλά αν σκεφτεί κανείς ένα θύμα, ότι αυτό το, αυτό το θύμα πρέπει να περάσει από συνεντεύξεις, από ανακρίσεις, πολλές φορές δεν, δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες και έτσι δεν πιστεύουν πολλές φορές τους ανθρώπους, τα θύματα. Και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχουν οργανώσεις που θα υποστηρίζουν τα θύματα, ιδίως τα ανήλικα θύματα. Για να συνοψίσω, η οδηγία προβλέπει λοιπόν τη συμμετοχή, την ενεργή των οργανώσεων, των υποστηρικτικών. Αυτές οι οργανώσεις πρέπει να μας βοηθήσουν να μάθουμε και τι είδους εκπαίδευση χρειάζονται ή το προσωπικό, χρειάζεται το προσωπικό των επίσημων αρχών. Επίσης για την ταυτοποίηση. Η ταυτοποίηση είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Δυστυχώ διαπιστώνουμε ότι πολλέ φορέ οι αστυνομικέ αρχέ ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έρχεται σε μια πρώτη επαφή με ένα θύμα, όπω είναι ένα νοσοκομείο για πράγμα. δεν έχει τι γνώσει για να προβεί στην ταυτοποίηση του θύματο. Γι' αυτό και χρειάζεται να δούμε πώ ακριβώ γίνονται οι συνεντεύξει, ιδίω με τα παιδιά. Και εδώ βλέπετε και στην έκθεση ότι έχουμε ξεχωριστό κεφάλαιο για τα παιδιά. Πρέπει να βρούμε τρόπου ώστε να μην ξαναζήσουν τα ίδια, να μην τραυματιστούν, να μην πληγωθούν ακόμα περισσότερο, ενώ είναι ήδη θύματα. Μιλάμε και για το φίλο του συνεντευξιάζοντος, αυτού που κάνει τη συνέντευξη. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα για να, ξεκαθαρι... για να εξασφαλιστεί ότι αυτή η διαδικασία της ταυτοποίησης θα γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο ώστε πραγματικά να παρέχει υποστήριξη προς το θύμα. Μιλήσαμε για ειδικέ ανάγκες, μιλήσαμε για διαταραχές, ε, ψυχικής υγείας, εγκυμοσύνες. Πολλές από τις γυναίκες που είναι θύματα τράφικινγκ μένουν έγκυες. Εκεί χρειάζεται να δοθεί μια ειδική υποστήριξη. Οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων. Βοηθάει, γιατί καθοδηγεί τα κράτη-μέλη στο πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους περιπτώσεις, τέτοιου είδους περιστατικά. Ψυχολογικά, υλικά, όλα αυτά είναι υποχρεώσεις. Δεν μπορεί κανείς να τις αποφύγει. Επίσης, μιλήσαμε για, μιλάμε για υποστηρικτικές υπηρεσίες στα κέντρα υποδοχής παιδιών και ανηλίκων. Όταν μιλάμε για κορίτσια δηλαδή που είναι κατά κύριο λόγο θύματα τράφικινγκ. Βλέπουμε σε, πολλά, σε πολλές χώρες τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τα υποστηρικτικά κέντρα τους. Αλλά για παιδιά που έχουν ε, δυστυχώς εκτεθεί σε τέτοιες αποτρόπιες εμπειρίες δεν αρκεί να τα στηβάζεις στα συνήθη κέντρα. Χρειάζεται λοιπόν να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν ειδική εξειδικευμένη υποστήριξη προς τα παιδιά που έχουν εκτεθεί σε τέτοιες αποτρόπες εμπειρίες. Επίσης, καθώς το τράφικινγκ για σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελεί μορφή έμφυλης βίας. Είναι σημαντικό να εξεταστεί και ξεχωριστά. Δεν είναι απλά άλλη μία μορφή του τράφικινγκ. Είναι μορφή βίας κατά των γυναικών. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι τα κράτη-μέλη ή πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμη στρατηγική για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Ή ακόμη και αν υπάρχουν, δεν προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση του τράφικινγκ. Γι' αυτό και εμείς συστήνουμε στις στρατηγικές αυτές, τις ολοκληρωμένες στρατηγικές για την ισότητα των φύλων, πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθούν σε κάθε κράτος μέλος μέτρα για την καταπολέμηση του τράφικινγκ. Ταυτοποίηση. Εμείς εκπονήσαμε μια μελέτη για το κόστος της βίας κατά των γυναικών και πρόκειται για τεράστιο κόστος, πρέπει να σας πω, που δεν θα έπρεπε να το επομίζονται οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αν προέβαιναν, δεν θα χρειαζόταν να το επομίζονται, αν προέβαιναν σε πρόληψη και δεν μιλάμε μόνο για, για την ε, εξασφάλιση της προστασίας των γυναικών, θα, που είναι το προφανές, θα βοηθούσε η πρόληψη στην εξοικονόμηση πόρων. βλέπουμε από τη μελέτη που κάναμε ότι ένας από τους λόγους για τον οποίο μπορεί ένα κορίτσι να διοικηθεί σε αναγκαστικό γάμο είναι η φτώχεια. Γιατί με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια του κοριτσιού παίρνει χρήματα. Αυτό αφορά και τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, όπως είναι η Ρωμά για παράδειγμα. Ακριβώς λοιπόν αν τα λάβουμε όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη μας μπορούμε να διαμορφώσουμε τις στρατηγικέ μας με, με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται όλοι οι κίνδυνοι. Υπάρχει και η πρωτοβουλία για την αστυνόμευση στις τοπικές κοινωνίες. Μιλήσαμε χθες με εκπροσώπους των ρουμανικών αρχών και μας είπαν ότι αυτός, αυτές οι περιπολίες οι τοπικές θα μπορούσαν να είναι ένας τρόπος πρόληψης για να μην αυξάνεται τουλάχιστον ο αριθμός και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου γιατί όχι και να μειωθεί επιτέλους αυτός ο αριθμός. Δικαιοσύνη και πρόσβαση των θυμάτων σε αυτή. Στην έκθεσή μας έχουμε εντάξει ένα σχετικό κεφάλαιο. Τα περισσότερα θύματα τράφικινγκ, κορίτσια και γυναίκες, Βεβαίω, όπω καταλαβαίνετε, δεν τους έχει μείνει ίχνος αυτοπεποίθηση. Βρίσκονται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και πολλές φορές δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στους, ε, στους θεσμούς της Είναι φοβισμένες και αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα εξαιτίας των εμπειριών τους. Βλέπουμε όμως ότι αν οι υπάλληλοι των φορέων αυτών, των εισαγγελικών αρχών, των δικαστικών αρχών, έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δυστυχώς η, η, αριθμή είναι πολύ χαμηλή. Τα, τα επίπεδα εκπαίδευσης είναι πολύ χαμηλά. Πολύ, πολλές φορές βλέπουμε δικαστές να μην πιστεύουν ή να μην δίνουν πολύ μεγάλη αξία. Ε, κάποιες φορές μέχρι και ο ο θήτης ε, παρεμβαίνει παρουσία του θύματος σε, σε παρεμβάσεις. Χρειάζεται βεβαίως ίση μεταχείριση, όμως χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη για τα θύματα. Στερεοτυπική πρέπει πραγματικά να κάνουμε ό,τι, ό,τι περνά από το χέρι μας για να ε, καταπολεμήσουμε στερεότυπα, όπως για παράδειγμα ότι πήγαινε γυρεύοντας και τέτοια. Όπω είπε και η Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών, χρειάζεται πραγματικά να υπάρξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η ισότητα των φύλων θα πρέπει να είναι στοιχείο που θα λαμβάνεται υπόψη πάντοτε και παντού. Εμείς λοιπόν καταλήξαμε και προτείνουμε σε εσά κάποιους δείκτες που θα μπορούσαν στο μέλλον με την αξιοποίηση των κατάλληλων στατιστικών δεδομένων να μας προσφέρει εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα εξαιρετικό εργαλείο για να παρακολουθούμε την κατάσταση και αναλόγως των επόμενων βημάτων που θα αναλυφθούν βεβαίως κάτι, τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους τους επαγγελματίες πρέπει να γίνει σήμερα. Σήμερα. Γιατί χάνουμε ζωές καθημερινά λόγω της έλλειψης γνώσεων και κατάρτισης. Σήμερα λοιπόν που είναι μέρα καταπολέμησης του τράφικινγκ είναι πραγματικά σημαντικότατο να προβούμε σε αυτές τις ενέργειες για να έχουμε και κάτι απτό να επιδείξουμε στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο των, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Thank you very much for giving me the floor and also it's such a pleasure. Χαίρομαι που είμαι μεταξύ σας σήμερα. Πράγματι είναι μια σημαντική ημέρα για την αναγνώριση του τράφικινγκ και για τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να εκριζωθεί αυτή η φρικτή πρακτική. Θέλω να συγχαρώ επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας για τη δημοσίευση αυτής της ιδιαίτερα εύθετης χρονικά έκθεσης για το τράφικινγκ. Θα ήθελα επίσης να θέσω τρία θέματα σχετικά με τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Όπως είπατε, πρέπει να έχουμε σωστά στοιχεία για να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Όπως λέει και το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ότι οι γυναίκες και τα παιδιά είναι το 70% των θυμάτων του ε, ε, τράφικινγκ, ιδιαίτερα στον τομέα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Υπάρχουν και άλλες πρακτικές σχετικά με το φύλλο που περιλαμβάνουν την καλύτερη διαδικασία ανείχνευσης των ε, γυναικών, όπως επίσης και το θέμα της προβληματικής των φύλων. Επίσης και το θέμα της ιδιότητας κάθε φορά του φίλου και του ρόλου που παίζει η ιδιότητα αυτή. Η δημοσίευση θα διευκολύνει, θα έλεγα, την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι μια βασική θεμελιώδης προτεραιότητα της ατζέντα για τα Ηνωμένα Έθνη. Θα πρέπει και η συνεργασία ανάμεσα στα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχιστεί και στα πλαίσια του λεγόμενου Glow Act ε, που εφαρμόζεται και από τα Ηνωμένα Έθνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το IOM, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. ιδιαίτερα και στον τομέα της προστασίας ε, και της φροντίδας των θυμάτων του τράφικινγκ. Έχει ξεκινήσει όπως ξέρετε και μια ενημερωτική εκστρατεία η οποία λέγεται My Story, Our Story και που περιγράφει θέματα σχετικά με τη βία εις βάρος των γυναικών. Υπάρχει και συλλογή μαρτυριών ε, και ε, εις βάρος ε, περιπτώσεων εις βάρος ανηλίκων και ενηλίκων. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα που να διασφαλίσουν την ειρήνη και την ασφάλεια. Ξέρετε ότι το τελευταίο βραβείο Νόμπελ δόθηκε στην Άντια Μοράντα. Είναι μια αναγνώριση του αγώνα τον οποίο έχει δώσει, ε, του αγώνα τον οποίο έχει δώσει η κυρία Μοράντα αναγνωρίζοντας ε, τη σημασία του προβλήματος. Η προσπάθεια ε, ανθρώπων που επιβίωσαν αυτής της απαράδεκτης πρακτικής όπως της κυρίας Μοράντ θα πρέπει να υποστηριχθεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για μια ακόμη φορά για την δημοσίευσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στις ερωταπαντήσεις. Κυρία Μπιόρκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και τις δύο προέδρους, τους δύο προέδρους των Επιτροπών, τους προσκεκλισμένους μας, την κυρία Βασιλιάδου και όλους όσους συμμετείχαν στην σύνταξη αυτής της έκθεσης. Με απασχολεί το θέμα αυτό. Ξέρετε ότι εμείς ως Κοινοβούλιο έχουμε ζητήσει στρατηγική για την καταπολέμηση του τράφικινγκ. Δυστυχώς δεν την έχουμε λάβει και αυτό είναι πραγματικά αξιολύπητο. Ε, το έχουμε ξαναπεί, εμείς το έχουμε ζητήσει, δυστυχώς όμως η Κομισιόν δεν μας έχει κάνει τη χάρη. Τράφικινγκ. όπως περιγράφεται στο έγγραφο που δημοσιεύτηκε πέρσι. Προφανώς υπάρχουν μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες Αφετέρου όμως υπάρχει αυτή η διολίσθηση να συνδεθεί το, το τράφικινγκ με την προσφυγιά και τη μετανάστευση. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί ξαφνικά ξεκινάει η συζήτηση ε, και πηγαίνει σε μια τελείως διαφορετική ε, κατεύθυνση. Προσπαθούν να την εκμεταλλευτούν διάφορες ε, δυνάμεις πολιτικές και κοινωνικές οι οποίες προσπαθούν να, να, να συνδέσουν τα πάντα όλα τα προβλήματα με τη μετανάστευση. Γι' αυτό Χαίρομαι που έχουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση που αναδεικνύονται οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος του τράφικινγκ, που μιλάμε για τα θύματα και που μιλάμε και για τους θύτες. Χαίρομαι που μιλάμε για τις αρχές επιβολής του νόμου, για μέτρα προφύλαξης και προστασίας και, προ... και πρόληψης. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ποια είναι η θέση μου. Από μία άποψη, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει. Πρώτον, να ξεριζώσουμε τη ζήτηση, να μειώσουμε και συνέχεια να εξαλείψουμε τη ζέστη ζήτηση. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το τράφικινγκ στις περισσότερες περιπτώσεις, στις πλήσεις περιπτώσεις καταλήγει σε σεξουαλική εκμετάλλευση. Γι' αυτό γίνεται. Γι' αυτό και πρέπει να μιλήσουμε για τις, αγοράς, για τις αγορές της πορνείας στην Ευρώπη. Και εκεί βλέπουμε ότι όπου υπάρχει μεγάλη αγορά πορνείας υπάρχουν και πάρα πολλά θύματα τράφικινγκ. Τα οποία βεβαίως θύματα καταλήγουν σε να, να πολλούνται σε αυτές τις αγορές της πορνείας. Ξέρουμε ότι στις δύο χώρες που έχουν θεσμοθετήσει την πορνεία παρατηρούμε αυτά τα φαινόμενα της αύξησης των, των θυμάτων του τράφικινγκ. Γιατί αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Εντάξει, μπορεί κάποιος να πει ότι δεν θέλουμε να επιτεθούμε στους 20 ανοχής για παράδειγμα κτλ, Φυσικά και είναι δύσκολο, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Φυσικά και είναι δύσκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το κάνουμε. Εμείς ως φεμινίστρες, ως φεμινιστές πρέπει να το κάνουμε. Ότι αυτό... Και να πούμε ξεκάθαρα ότι εδώ δεν μιλάμε για σεξουαλική ελευθερία. Μιλάμε για, για καταπίεση σεξουαλική και για εκμετάλλευση ε, αδυναμιών ε, ιερόδουλες, ε, προαγωγή. Όλα αυτά πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους. Υπάρχουν εκείνοι που πουλάνε και εκείνοι που αγοράζουν αυτές οι υπηρεσίες. Εγώ ξέρετε είμαι Σκανδιναβή. Αλλά είναι σαφές για μένα ότι πρέπει να τιμωρούνται, να ποινικοποιούνται και εκείνοι που αποδέχονται υπηρεσίες από θύματα τράφικινγκ. Είναι υποχρέωσή τους να μάθουν ποιος είναι αυτός που τους προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, θα, θέλα, θα ήθελα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δούμε πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε τις διοκτικές αρχές, πώς οι εισαγγελικές αρχές, οι ανακριτικές αρχές, οι αστυνομικές αρχές θα μπορούσαν να, να συνεργαστούν, να συλλέγουν όλες τις, δυνατό, τις δυνατές πληροφορίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Υπάρχουν δίκτυα, υπάρχουν και χώρε που έχουν διανύσει ήδη αυτό το δρόμο, που τον έχουν χαράξει. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που δεν, που δεν τον έχουν διανύσει, που δεν έχουν φτάσει πολύ μπροστά, αλλά μπορούν να υπάρξει, μπορεί να υπάρξει μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει πολύ μεγαλύτερη δράση. Εμείς είμαστε... <coughs> Είμαστε παράγοντα έλξη. Βεβαίω, εδώ υπάρχει ζήτηση. Αυτό δημιουργεί και την υποχρέωση να ερευνήσουμε ε, τις υποθέσεις αυτές, να κρατήσουμε τα κορίτσια στο σχολείο. Ε, ο μέσος όρος ηλικίας ποιος είναι, 16 χρονών αυτών των κοριτσιών. Ε, το βασικό είναι να κρατήσουμε τα κορίτσια στο σχολείο και θα μειωθεί ο αριθμός των θυμάτων σωματιμπορίες. Ε, είμαστε πολύ καλύτεροι, ε, γιατί δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στη διάσταση του φύλου, αλλά πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα και ένα από αυτά είναι να σταματήσουμε την ατιμορρησία και να ε, εστιάσουμε σε αυτό που λειτουργεί, δηλαδή στη μείωση της ζήτησης. Η κυρία Κινίτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους α, ε, ομιλητές μας για τη δουλειά που έκαναν, για την παρουσίαση που έκαναν, για το θέμα αυτό που είναι τόσο σημαντικό η σωματεμπορία που τη διαχειρίζονται εγκληματικές οργανώσεις και σε διεθνές επίπεδο. Συμφωνώ με αυτά που είπατε ότι κυρίως γίνεται για να εκμεταλλευτούν σεξουαλικά αυτά τα άτομα. Συνήθως αφορά τις γυναίκες, αλλά και πολλούς ανηλίκους και κυρίως κορίτσια. Δεν είναι μόνο μια μορφή βίας ειδική έμφυλη βία, αλλά πάνω απ' όλα είναι μια παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πώ θα την αντιμετωπίσουμε, πώ θα την καταπολεμήσουμε, με το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. Πάνω απ' όλα, πιστεύω εγώ. Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ σε αυτή την οδηγία που μιλήσατε για την ε, σωματεμπορία και την ε, οδηγία για τα θύματα. Θα πρέπει να εφαρμοστούν συντονισμένα και οι δύο δηλαδή οδηγίες. Και εγώ πιστεύω ότι ορισμένες χώρες πρέπει να κάνουν πολλά ακόμη, ούτως ώστε να εφαρμόσουν σωστά αυτές τις οδηγίες. Ε, ακούστηκαν και άλλες σκέψεις από τους ομιλητές μας, αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε, να παρακινήσουμε τα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν τις δύο οδηγίες. Ο ρόλος της Europol είναι σημαντικός για αυτά τα θέματα σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και το συντονισμό κυρίως. Μήπως θα μπορούσαμε αυτό το ρόλο να τον ενισχύσουμε ακόμα περαιτέρω, τρόπος της ε, Europol και κυρίως ε, μήπως θα μπορούσε να συντονίζει τις ε, δράσεις των διαφόρων διοκτικών αρχών. Αυτή η δραστηριότητα συνεργασίας δηλαδή είναι πολύ σημαντική και είναι εργαλείο για συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε και σε διεθνές επίπεδο τους διακινητές ανθρωπίνων όντων. Ένα άλλο στοιχείο που κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σημαντικό και εγώ έχω ασχοληθεί και στο παρελθόν στο Κοινοβούλιο είναι το θέμα της ε, προστασίας των ανηλίκων. Η προστασία των θυμάτων γενικά είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα. Ε, δίκαιο και δικαιοσύνη. Με αυτά τα εργαλεία καταπολεμούμε την ε, εμπορία ανθρώπων. Αλλά θα πρέπει να πλαισιωθεί όλο αυτό από συγκεκριμένα μέτρα, μέσα στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματο υπέρ των θυμάτων, για τη στήριξη των θυμάτων, για τη βοήθεια των θυμάτων. Ε, σε μια πρώτη φάση, ε, όπω υπόθηκε σωστά, είναι το θέμα είναι να, ταυτο, να ταυτοποιήσουμε τα θύματα, τους ε, ενεχόμενους. Θα πρέπει οι αστυνομικέ αρχές να κάνουν αυτή τη δουλειά, να συνεργαστούν, γιατί είναι το front office, ας πούμε, για να αντιμετωπίσουν τα θύματα αυτών των αδικημάτων. Εγώ προσωπικά πιστεύω, πιστεύετε κι εσείς ότι θα πρέπει να κάνουν περισσότερες προσπάθειες για να καταρτήσουμε τους αστυνομικούς. Τι λέτε γι' αυτό. Και ένα άλλο στοιχείο, στη χώρα μου την Ιταλία δημιουργήθηκε ένα πραγματικό σύστημα στήριξης των θυμάτων με παρουσία από τις τοπικές αρχές, από υγειονομικές αρχές, από εκπροσώπους, από οργανώσεις. Γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά και κορίτσια, για κοριτσάκια πολύ μικρά, να υπάρχει μία πολύ λεπτή προσέγγιση. Και για να δούμε τι απασχολεί τα θύματα, πόσο υπέφεραν, πού υπέφεραν, αλλά και για να ε, υιοθετήσουμε τα κατάλληλα μέτρα για να τις βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τα τραύματά τους, παρότι δεν είναι εύκολο. Εσείς πιστεύετε, λοιπόν, ότι πρέπει να υπάρχει ένα κανονικό, ολοκληρωμένο σύστημα στήριξης των θυμάτων. Αυτά και σας ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος θα έρθει όπου να είναι. Έτσι μου είπανε. Η κυρία Σίπελ, θα ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ καταρχάς που ε, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να σας πω ότι ντρέπομαι. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Είμαστε στον 21ο αιώνα και η κυρία ε, Βασιλιάδου μόλις μας ενημερώσε ότι ο αριθμός των θυμάτων εδώ στην Ευρώπη αυξάνεται. Με σοκάρει πραγματικά το γεγονός αυτό. Και με σοκάρει το γεγονός ότι η συζήτηση επικεντρώνεται στο τράφικινγκ και ε, στη μετανάστευση. Ενώ αυτό που θα έπρεπε να συζητάμε είναι η ζήτηση. Και με ανησυχεί ε, το γεγονός ότι δυστυχώς έτσι με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζουν και οι ιδιοκτικές αρχές των κρατών μελών το θέμα. Δεν πιστεύω ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορούμε να το καταπολεμήσουμε, να το αντιμετωπίσουμε με, το, με την καταπολέμηση των εγκληματιών. Και μόνο. Η κυρία Βασιλιάδου είπε, αν εξαλείψουμε το κέρδος, λύνεται το πρόβλημα. Δυστυχώς φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Διότι Υπάρχουν δύο όψει του νομίσματος. Αφενό είναι η εγκληματικότητα, οι, εγκλημα... οι εγκληματίες και από την άλλη πλευρά υπάρχει και η φτώχεια. Φυσικά ενδέχεται κάποια στιγμή ε, και κορίτσια από πιο πλούσιε οικογένειε να γίνουν θύματα, Όμω η αλήθεια είναι ότι όσο, μεγαλύτερο, όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνο τη φτώχεια που αντιμετωπίζει ε, μια οικογένεια με τα κορίτσια τη τόσο μεγαλύτερο είναι ο κίνδυνο, τελικά τα παιδιά του να γίνουν ε, θύματα του τράφικινγκ. Έχω και μια ανησυχία ε, σε σχέση με το εξή. Πού τελικά συμβαίνει αυτή η κακοποίηση. Μιλάμε πάρα πολύ για το ίντερνετ. Και εντάξει, εν μέρη, αν παρακολουθούμε βεβαίως τις φωτογραφίες και ποιο τελικά τις βάζει στο δίκτυο κτλ. Μπορεί να βοηθούν όλα αυτά να βρούμε ε, τα, τους Ξεχνάμε όμως ότι πίσω από κάθε φωτογραφία, πίσω από κάθε βίντεο υπάρχει μια σεξουαλική κατοποίηση η οποία συνέβη στην πραγματική ζωή. Αναρωτιέμαι λοιπόν, δεν γνωρίζουμε πότε εξαφανίζεται μια γυναίκα, πότε εξαφανίζεται ένα κορίτσι, πότε αρχίζει μια γυναίκα ή ένα κορίτσι να συμπεριφέρεται διαφορετικά. Εδώ υπάρχει τεράστιο καθήκον που αφορά όχι μόνο τις αστυνομικές δικαστικές αρχές, αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Όταν και εδώ στο Κοινοβούλιο μιλάμε για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, υπάρχουν συνάδελφοι που ισχυρίζονται ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να μιλάμε μόνο για τη βία κατά των γυναικών, αφού ασκείται βία και κατά ε, ε, άλλων πληθυσμιακών ομάδων, κοινωνικών στρωμάτων. Το βρίσκω πραγματικά σοκαριστικό, ντροπιαστικό. Οι γυναίκες είναι το 50% του πληθυσμού, εδώ και αιώνες καταπιέζονται. Το γεγονός ότι δηλαδή καλούμαστε ακόμη σήμερα να λέμε τα αυτονόητα αποδεικνύει πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. <clears throat> Γι' αυτό και ελπίζω με όλους τους ε, εταίρους μας να καταφέρουμε, να καταφέρουμε επιτέλους να χαράξουμε, να δημιουργήσουμε μια στρατηγική ώστε τα επόμενα χρόνια να σταματήσουμε να ακούμε ε, αυτές τις πολύ ε, ε, λυπηρές ε, ειδήσει για αύξηση των θυμάτων. Ευχαριστώ. Μαχτά, στο τέλος. Ευχαριστώ. Ε, άκουσα με μεγάλη προσοχή τις παρουσιάσεις, τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Εγώ είμαι από εκείνου που συνδέουν την φτώχεια με τη σωματεμπορία φυσικά. Αλλά δεν υπάρχει μόνο αυτή η διάσταση. Παρότι υπάρχει έντονα, υπάρχουν οικογένειες ε, που παντρεύουν ε, τις ανήλικες κόρες τους γιατί δεν έχουν λεφτά. Το είπατε κυρία μου και είναι μια πραγματικότητα, θα, δούμε, θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, να την καταπολεμήσουμε. Πέρυσι είχα πάει στη Σικελία. Εκεί από εκεί περνάνε πολλές γυναίκες ε, και γυναίκες από τρίτες χώρες, αλλά και Ευρωπαίες. Ε, Ρουμάνες διακινούνται μέσω της Σικελίας. Εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι η δικαιοσύνη έχει πολύ λίγα μέσα στη διάθεσή της. Ε, η εισαγγελία είναι μόνη τη, με τρία άτομα, με τρει βοηθού για να καλύψει όλη τη συγκελία. Φυσικά υπάρχουν οργανώσει που αναλαμβάνουν τα θύματα, αλλά είναι εντελώ ανεπαρκέ αυτό το επίπεδο. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για την Ισπανία, για τη Βουλγαρία, για τη Ρουμανία, ακόμα και για το Βέλγιο και για τη Γαλλία, για τη Γερμανία. Εγώ είμαι σε μια συνοριακή περιοχή της Γαλλίας δίπλα στην ε, Γερμανία. Λίγα χιλιόμετρα από το σπίτι μου υπάρχει το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος οίκος ανοχής της Ευρώπης. Πάνω από χίλιες ιερόδουλες ε, προϊόν όλων των ειδών σε ματεμπορία, σε σεξουαλικής εκμετάλλευσης και γυναίκες σε μεγάλη πλειοψηφία ανήλικες. Τα ξέρουν όλοι. Όλοι τα ξέρουν αυτά. Εγώ ξεκινάω από την αρχή ότι αν η Ευρώπη θέλει να καταλήψει αυτήν την υποκρισία και να, κάνει, να το κάνει μπαντιέρα ευρωπαϊκή, να καταπολεμήσει την πορνεία και τη σωματεμπορία. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, δικαιωμάτων των γυναικών, δικαιωμάτων των προσώπων. Θα πρέπει καταρχάς να εναρμονίσουμε τις νομοθεσίες μας για το θέμα της πορνείας. Γιατί υπάρχουν χώρες όπου απαγορεύεται, σε άλλες που είναι νόμιμη, σε άλλες που την ανεχόμαστε κτλ. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Αλλά για να μην ακρηγορήσω, για να τελειώσω. Ωραία. Εγώ Θέλω όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όλοι και όλες, να πούμε ότι θα γίνει η ευρωπαϊκή πανδιέρα. Πανδιέρα η καταπολέμηση της πορνείας και του εθεμπορίου ανθρώπων. Από όπου και αν προέρχεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, δίνει περισσότερα μέσα στη Frontex, γιατί θεωρεί έτσι, και ο καθένα θα το εκτιμήσει αυτό, ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση κυρίως. Ποια είναι τα μέσα σήμερα που δίνουμε στα διάφορα, στους διάφορους θεσμούς, ε, στις αστυνομικές αρχές, στις διάφορες οργανώσεις για να καταπολέμησουν αυτή τη μάστιγα. Τι λεφτά τους δίνουμε. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να φτιάξουμε ένα αντίστοιχο Frontex για να καταπολεμήσουμε τη σωματεμπορία. Δεν υπάρχει κάτι το αντίστοιχο. Χρειάζονται και λόγια αλλά και πράξεις πάνω απ' όλα, έτσι. Ωραία. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Έχουμε τον κύριο Επίτροπο μαζί μας. Μιλάμε για τα ειδικά μέτρα στα πλαίσια της καταπολέμησης του τράφικινγκ, τα οποία διέπονται από την προβληματική των φύλων. Έχει ολοκληρωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα μέλη. Τώρα θα ακούσουμε ε, με ικανοποίηση τις παρατηρήσεις σας. Πρόεδρε, συνάδελφοι, αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσω λέγοντας ότι λυπάμαι γιατί ήμουν απόν. Ξέρετε όμως ότι είναι μια δύσκολη μέρα για μένα. Έρχομαι απευθείας από την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού και την διαδικασία απαλλαγής. Η μέρα λοιπόν σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, είναι η μέρα εναντίον του τράφικινγκ για την Ευρώπη. Η μέρα αυτή μας υπενθυμίζει σε όλους ε, τις συλλογικέ μας ευθύνες να συνεχίσουμε και να βελτιώσουμε τις προσπάθειές μας ε, για να εκριζώσουμε αυτό το μισητό έγκλημα, να στηρίξουμε κάθε θύμα και θα πρέπει επίσης να, ε, να θυμόμαστε αυτήν την μέρα, όχι μόνο σήμερα, αλλά σε καθημερινή βάση. Το τράφικινγκ, η σωματεμπορία, εν πάση περιπτώσει, δεν διεξάγεται μόνο στη Λιβύη, όπως κάποιοι πιστεύουν, ή σε κάποιες άλλες περιοχές μακράν της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά διεξάγεται και εντός των ευρωπαϊκών μας κοινωνιών. Είναι κάτι το οποίο όλοι συνειδητοποιούμε ενστικτοδός, αλλά έχουμε και στοιχεία πλέον για να το τεκμηριώσουμε. Πρόκειται για το έγκλημα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών κυρίως και νέων κοριτσιών. Από την πρώτη στιγμή ε, που ανέλαβαν τις ευθύνες ε, του χαρτοφυλακίου μου εδώ και τέσσερα έτη, συμπεριλαμβάνεται σε αυτές ε, και η καταπολέμηση του τράφικινγκ, εγώ ζήτησα να υπάρξουν απτά αποτελέσματα και συγκεκριμένα κατορθώματα, αν θέλετε. Ο μόνος τρόπος ε, είναι η συνεργασία με τα κράτη-μέλη, με τα ευρωπαϊκά όργανα και φυσικά με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, όπως το κάνουμε σήμερα μέσω αυτής εδώ της ε, συναντήσεως. Εσείς, τα μέλη των Επιτροπών ΦΕΜ και ΛΥΜΠΕ, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, όπως επίσης και η συντονίστριά μας μάλλον για τα θέματα καταπολέμησης του τράφικινγκ, ο συντονισμός και η συλλογική δράση είναι καθοριστική για την επιτυχία της πολιτικής μας στον τομέα του τράφικινγκ. Η έκθεση για τα ειδικά μέτρα με ε, λήψη υπόψη του φύλου μας δίνει την δυνατότητα να συζητήσουμε κάποιες βασικές ε, απτές προτεραιότητες. Εγώ παρουσίασα το Δεκέμβριο του 2017 μέτρα έτσι ώστε να προχωρήσουμε με στοχευμένο και συγκεκριμένο τρόπο τα μέσα καταπολέμησης του τράφικινγκ. Η έκθεση ε, έχει σαν στόχο να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να σεβαστούν, να φέρουν εις πέραν τις υποχρεώσεις τους, πέρα στις υποχρεώσεις τους, υιοθετώντα μέτρα τα οποία να εμπνέονται από την προβληματική του φύλου. Συνεισφέρει η έκθεση αυτή τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε για την υποστήριξη των μέσων αυτών και την στήριξη επίσης ε, των ε, θυμάτων. Αλλά δεν μιλάμε μόνο για γυναίκες, υπάρχουν και πάρα πολλοί ανήλικοι άνδρες, ε, αγόρια που γίνονται, που πέφτουν αντικείμενα, συγγνώμη, που τους εκμεταλλεύεται η εγκληματική αυτή πρακτική. Ε, υπάρχουν ε, εγκληματικά δίκτυα ε, τα οποία ασκούν αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες, δράσεις και εκμεταλλεύονται τους ανηλίκους. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πετύχει κάποιους πρώτους στόχους, τα θύματα δηλαδή του τράφικινγκ να υποστηριχθούν και τα δικαιώματά τους να προστατευθούν. Πριν το τέλος του χρόνου θα ξεκινήσω επίσης και την δεύτερη έκθεση καταπολέμησης του τράφικινγκ. Θα παρουσιάσουμε ε, νέα μέτρα και θα καταμετρήσουμε, θα αξιολογήσουμε την εφαρμογή των μέτρων μέχρι σήμερα. Ε, σήμερα την ημέρα λοιπόν καταπολέμησης ε, της, ε, του τράφικινγκ στην Ευρώπη και παγκόσμια σας ζητώ από όλους να ενώσετε τις δυνάμεις σας και να πάρετε μέρος στις προσπάθειές μας. Να σταματήσουμε, να τερματίσουμε κάθε μορφή εκμετάλλευσης, να αντιμετωπίσουμε τα θύματα με την αξιοπρέπεια που τους οφείλουμε. Να έχουμε μηδενική ανοχή απέναντι στην κουλτούρα της ατιμορρησίας και κυρίως να αποτρέψουμε να πέσουν και άλλοι άνθρωποι θύματα αυτής της πρακτικής. Το τράφικινγκ των γυναικών και των κοριτσιών είναι κάτι το οποίο είναι αντίθετο με την ισότητα που μας εμπνέει, με την αξιοπρέπεια που πρέπει να χαρακτηρίζει τη ζωή όλων. Δεν υπάρχει θέση για το τράφικινγκ και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και ουδήποτε αλλού στον κόσμο. Έχουμε λοιπόν το ηθικό καθήκον να προχωρήσουμε στη λήψη μέτρων και να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, να ξεφύγουμε πια από τα λόγια. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να δώσω το λόγο στους ομιλητές μας τώρα για να απαντήσουν ε, εν συντομία στις ερωτήσει και τι παρατηρήσει που ακούστηκαν. Δύο λεπτά σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Όλα τα σχόλια θεωρώ ότι σχετίζονται με τη συνολική εικόνα, την εναρμόνιση των, ε, της νομοθεσίας που απαιτείται. Και νομίζω ότι ένας από τους τρόπους που μπορεί κανείς να προσεγγίσει το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές εθνικές, ε, υπάρχουν πάρα πολλές νομικές πράξεις. Υπόθηκε από πολλούς ότι το θέμα είναι η ζήτηση. Δυστυχώς όμως ε, το θέμα προσεγγίζεται διαφορετικά στα, στα κράτη-μέλη. Ούτε, ούτε συγκριτικά στοιχεία δεν μπορούμε ε, να, να εξάγουμε αξιόπιστα πόσο μάλλον ε, τις διάφορες αρχές, τις διάφορες υπηρεσίες, τους διάφορους μεθόδους προσέγγισης, αντιμετώπισης του προβλήματος. Οπότε η σημαντικότερη δυνατότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η μείωση της ζήτησης. Αναφέρθηκε και η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Τα σχολεία λοιπόν, όχι μόνο οι αστυνομικέ αρχές, και τα σχολεία έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των παιδιών που, και των κοριτσιών κυρίως που, που ε, κινδυνεύουν. Υπάρχουν λοιπόν πολλά περιθώρια βελτίωσης από την πλευρά των κρατών μελών όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αυτό συνδέεται με το πόσες πληροφορίες λαμβάνουν, τα, ακόμη και στο σχολείο, τα κορίτσια. Πόσο υποστηρίζουμε τις, ε, τις ευάλωτες ομάδες όπως είναι η Ρωμά ή τους μετανάστες που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη διαδικασία ένταξής τους στις κοινωνίες μας. Δεν μπορεί κανείς το, την καταπολέμηση του, του τράφικινγκ να την αναθέσει σε έναν και μόνο τομέα, στην αστυνομία για παράδειγμα ή στο δικαστικό σύστημα ή στο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να διαπνέει μια σειρά από τομείς η προσπάθεια αυτή, η επιδίωξη να καταπολεμηθεί το τράφικινγκ. Κυρία Βασιλιάδου, ευχαριστώ. Δεν έχω αλλά δεν χρειάζομαι και πολύ χρόνο γιατί νομίζω ότι η παρουσία του Επιτρόπου είναι εύγλωτη από μόνη της. Απλώς να απαντήσω σε, κάποια, σε κάποιες από τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Εμείς παρακολουθούμε στενά τις υποχρεώσει των κρατών μελών που απορρέουν από την οδηγία για την υποχρέωσή του να, μεταφέρουν τις διατάξεις της οδηγίας στο εθνικό του δίκαιο. Το ίδιο κάνει και η Κομισιόν. Εμείς έχουμε μια πολύ ολοκληρωμένη ε, προσέγγιση και τονίζουμε ότι η υπήκοη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα περισσότερα θύματα τράφικινγκ, οπότε συνδέεται με τη μετανάσταση, αλλά όχι μόνο με τη μετανάστευση. Θέλουμε πάρα πολύ να συνδυάσουμε, να εξασφαλίσουμε το ότι η χρηματοδότηση θα αντιστοιχεί στις προτεραιότητες πολιτικής μας και, και ένα από τα παραδείγματα ε, για να απαντήσω και σε Ευρωβουλευτή είναι ότι χρηματοδοτούμε και ε, εθνικά προγράμματα μέσω, μέσω της αστυνομίας ISF. Και αυτό, τέτοια προσήλωση έχει εκφραστεί και από πλευρά Κομισιόν. Προσφέρουμε χρηματοδότηση μέσω διαφόρων προγραμμάτων. Κλείνω με αυτό που είπε και ο Επίτροπος. με τις δράσεις που αναφέρονται και στην ανακοίνωση του 2017. Πρέπει να σταματήσει η κουλτούρα της ατιμορρησίας. Αυτό θα πρέπει να είναι σε τελική ανάλυση ο στόχος. Πρέπει να σταματήσουν οι ροές κεφαλαίων, να σταματήσουν οι ροές χρημάτων, να σταματήσει η εκμετάλλευση. Αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει στρατηγική. Δεν υπάρχει μεν στρατηγική, υπάρχουν όμως πολύ συγκεκριμένες επιχειρησιακές δράσεις, τις οποίες και περιγράψαμε εδώ. Είναι πολύ συγκεκριμένες, πολύ απτές, αποφέρουν αποτελέσματα και αυτές ακολουθούμε στη συνεργασία μας με τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας σήμερα εδώ και για την πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτησή σας. Ευχαριστώ όλους τους προσκεκλημένους ομιλητές μας. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Πιμέντα Λόπες για το ότι συμπροείδρευσε μαζί μου τις συνεδρίες αυτής. Άρθρο 23, παράγραφος 1, προβλέπει ότι θα εκδοθεί και ε, έκθεση προόδου και την περιμένουμε πριν από την εκπνοή της φετινής χρονιάς. Ωραία. Τελειώνουμε με αυτό το θέμα λοιπόν. Να ζητήσω από την Μπάρμπαρα Σπινέλη να με αντικαταστήσει για να περάσουμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.